I will use this one. Uh, so, uh, <clears throat> once again, we... Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε στο σημείο 1, έγκριση της μερίσιας διάταξης. Προτείνεται η εξής αλλαγή. Το σημείο 11 να συζητηθεί μετά το σημείο 7. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Ήθελα να σα ενημερώσω επίση ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνάντηση και οι χρονοθίδε είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν στη διάρκεια τη συνεδρίαση. Σε ό,τι αφορά το σημείο 2, ανακοινώσει του Προέδρου, θα ήθελα να σα ενημερώσω για τι αποφάσει των συντονιστών. Στη συνεδρίασή του στι 4 Μαρτίου έλαβαν οι συντονιστέ τι εξή αποφάσει να ζητήσουν καταρχάς από την διάσκεψη των Προέδρων να ολοκληρώσει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών φορσοδήματος από ορισμένε εκμεταλλεύσει και κλάδους παρατήματα. Είναι κοινό σφάγγελο έκον γιούρι μέσω απλουστευμένη διαδικασίας την Ολομέλεια του Μαρτίου, τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου Επίση, με γραπτή διαδικασία που ολοκληρώθηκε την εβδομάδα παριθμών 10, αποφάσισαν οι συντονιστέ να απαντήσουν στο ερώτημα 1 του κεφαλαίου 3 τμήμα Α και στην ερώτηση 1 του κεφαλαίου 3 τμήμα Β του ερωτηματολογίου για την 21η ξαμηνή έκθεση τη ΚΟΖΑ και να μην απαντήσουν τι άλλε ερωτήσει, διότι απευθύνονται στα κοινοβούλια συνολικά. Σημείο 3 Αν δεν λάβουμε αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίας, τα πρακτικά της συνεδρίας 19 Νοεμβρίου του 18, της 20 Φεβρουαρίου του 19 και της 26 Φεβρουαρίου του 19 θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Για το σημείο 4, επικουρικότητα, δεν έχουμε κάτι. Επομένως μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 παρουσίαση της μελέτης που ανατέθηκε από το θεματικό τμήμα ΓΑΜΑ με θέμα τη μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του οικογενειακού δικαίου. μελέτη πραγματεύεται την ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική συνεργασία μεταξύ Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου στην τομέα του γενικού δικαίου μετά το Brexit και πιο συγκεκριμένα εξετάζει τα διάφορα πιθανά νομικά σενάρια στο στάδιο της ε, αποχώρησης και της μελλοντικής σχέσης στον τομέα του γενικού δικαίου. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα ήθελα να καλωσορίσω δύο εμπειρογνώμονες της ομάδος ε, που συνέταξαν αυτή τη μελέτη, Μάρτα Ρεκέχο Ισίδρο, από το Μάξ Planck στο Λουξεμβούργο, ερευνήτρια και τον Τιμ Άμος, ε, δικηγόρο, από το Ηνωμένο Βασίλειο. 20 λεπτά έχετε και ίδιο στη διάθεσή σας. Παρακαλώ μοιραστείτε το χρόνο μεταξύ σας, όπως επίσης επιθυμείτε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Συμφωνήσαμε με την ε, κυρία Ρεκέχο Ισίδρο να ξεκινήσω εγώ αρχικά για να θέσω λίγο το πλαίσιο. Η έκθεση ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2018 και τώρα είμαστε 12 ημέρες πριν την λήξη προθεσμίας ε, για την αναξισχύωση του Brexit. Δεν έχουμε μέχρι στιγμή συμφωνία, άρα δεν έχουμε ούτε δίκαιο ούτε κάποια καθοδήγηση που ήταν μια από τις ε, τελικές συστάσεις της έκθεσης στη σελίδα 36. Εγώ βέβαια δεν μιλώ εδώ πολιτικά και το τονίζω αυτό, πάντως τα κατάσταση είναι κατεπίγουσα, είναι σοβαρή, ιδίω σε ό,τι αφορά τις οικογένειες και τα παιδιά που θα υποφέρουν μετά από 12 μέρες και μετά. Δικαιοδοσία, ποιο δικαστήριο θα ασχολείται με τι. Και αναγνώριση κυρίως των δικαστικών εντολών ή αμοιβαιότητα δηλαδή σεβασμός άλλων εντολών ε, και διαταγών και εκτελεστότητα αποφάσεων. Πραγματικά μιλάμε για ε, σημαντικά συστήματα οικογενειακού δικαίου. Εγώ δραστηριοποιούμαι στην Αγγλία και στην Ουαλία σε τέτοια θέματα ω δικηγόρο και προβλέπω ότι αν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο για το οικογενειακό δίκαιο και για αυτέ τι οικογένειε και αυτά τα παιδιά, θα έχουμε πραγματικά επίθεση κατά των πολιτικών από τους δημοσιογράφους ε, ένθεν κακήθεν της μάχης γιατί θα έχουν ε, αποτύχει πολιτική και θα έχουν απογοητεύσει ε, τις οικογένειες αυτές και τα παιδιά για τα επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια βέβαια δεν μιλάμε για επιχειρησιακό σχεδιασμό αλλά για οικογενειακό προγραμματισμό υπό την βασικότερη όμως έννοιά του, άρα οι τρεις επιλογές αναφέρονται στην έκθεση 24, το No Deal, δεύτερη επιλογή συνέχεια, Δηλαδή στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει να ισχύει μονομερό ε, η ενωσιακή νομοθεσία, αλλά αυτό δεν λειτουργεί λόγω έλλειψη ε, αμοιβότητας. Και τρίτη επιλογή είναι μια συμφωνία που φαίνεται πιθανή αλλά δεν είναι και τόσο σίγουρη. Thank you so much. Uh, in the study, we were asked to mm, address two sets of. Στην ε, μελέτη αυτή μας ζητήθηκε να εξετάσουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι το θέμα του χωρισμού, στην περίπτωση που υπάρχει συμφωνία, ε, αποχώρηση χωρίς συμφωνία, αλλά και αν υπάρξει και συμφωνία χωρίς να αποδίδεται σημασία σε το θέμα τόσο πλευράς ε, ευρωπαϊκή Ένωσης όσο και Ηνωμένου Βασιλείου. Και όπως είπε και ο Τιμ, ε, το επόμενο θέμα που ενδιαφέρει είναι οι προοπτικές κάποιες συμφωνίες και τι θα συμβεί στην περίπτωση μη συμφωνίας. Πριν λοιπόν μπούμε σε βάθος σε αυτά τα θέματα, θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τα πορίσματα της ε, μελέτης μας ε, που σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και αν η μελέτη προέκυψε τον Οκτώβριο που μας πέρασε και ορισμένα θέματα πρέπει να επικαιροποιηθούν. Στη μελέτη μας λοιπόν λέμε ότι για, τους, για τα μεμονωμένα άτομα η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη ε, στην περίπτωση βέβαια που υπάρχει μια συμφωνία αποχώρησης. Η μελέτη όμως εντοπίζει κάποιες ερμηνευτικές δυσκολίες αυτής της συμφωνίας ε, και αποδίδει σημασία και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που καλείται να ξεκαθαρίζει ορισμένα θέματα. Τώρα, κατά πόσον ε, θα υπάρξει συμφωνία αποχώρηση με συμφωνία ή όχι, όλοι εργάζονται μέσα σε ένα σχιζοφρενικό πλαίσιο όλοι προετοιμάζονται για αποχώρηση με συμφωνία, αλλά και για το αντίθετο σενάριο. Επίσης, η μελέτη καθιστά σαφές ότι υπάρχει αμοιβαιότητα, η ε, και οι δύο πλευρές θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όλοι επιβεβαιώνουν την ε, ε, αμοιβαιότητα, αλλά σε λιγότερο βαθμό. Μας ζήτησαν επίσης να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις του Brexit όσον αφορά την εναρμόνιση του οικογενειακού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει οθετήσει όλα τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει συμμετάσχει και σε όλες τις διαπραγματεύσεις. Οι δυσκολίες υπάρχουν στο οικογενειακό δίκαιο και αυτό οφείλεται κυρίω στι νομοθετικές διαδικασίε που είναι απαραίτητε λόγω του ότι το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο και ε, αυτό θα συνεχιστεί να υπάρχει ακόμα και αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην περίπτωση λοιπόν που υπάρξει συμφωνία, αποχώρηση με συμφωνία, που μάλλον ε, πιάζει, μοιάζει να συμφώνησαν από αυτού οι διαπραγματευτέ τον Νοέμβριο που μα πέρασε, θα έχουν μπροστά μα δύο χρονικέ περιόδου. Η πρώτη θα είναι μεταβατική περίοδο, η οποία θα αρχίσει την ημέρα αποχώρησης, κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί στις 31 ε, Δεκεμβρίου του 2020. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου θεωρούμε ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν ω έχουν, δηλαδή το ενωσιακό κεκτημένο θα ισχύει χωρίς καμία εξαίρεση και αυτό για οικογενειακά θέματα ε, σημαίνει ότι ε, θα διατηρηθούν όλοι οι κανονισμοί και ο 606 του 2003 που αφορά την προστασία σε αστικά θέματα. Ε, τώρα, όσον αφορά την περίπτωση που δεν υπάρξει η συμφωνια 6066 εως αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν από τον Ιανουάριο του 2021 και θα περιλαμβάνουν τις ε, διαδικασίες ε, που θα τρέχουν κατά το τέλος της μεταβατικής περίοδου και επίσης ε, και παράλληλες διαδικασίες θα ισχύει η δικαιοδοσία η οποία ε, θα εφαρμοστεί, η οποία θα αφορά τόσα τα νοσιακά δικαστήρια, όσο και τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά την αναγνώριση και την εφαρμογή, η διαδικασία η διατήρηση και οι δύο αυτά θα αρχίσουν να ισχύουν μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Εδώ ισχύουν τα έγγραφα τα οποία έχουν καταγραφεί ως αυθεντικά εργαλεία και συμφωνίες οι οποίες έχουν συναυθεί πριν από το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Όσον αφορά τώρα τη συνεργασία, οι ε, διαδικασίες που θα έχουν ζητηθεί από τις κεντρικές ή τις αρμόδιες αρχές πριν από το τέλος της μεταβατικής περίοδου, αυτές θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου με βάση τους ε, κανόνες ε, οι οποίοι θα έχουν θεσπιστεί. Όσον αφορά τα πισταποιητικά για προστατευτικά μέτρα, αν αυτά έχουν εκδοθεί πριν από το τέλος της μεταβατικής περίοδου, θα τεθούν σε ισχύ με βάση τον ενωσιακό κανόνα κανονισμό που ε, προβλέπει τι θα γίνει μετά τη μεταβατική περίοδο. Όπως σας ανακοίνωσα ήδη, υπάρχουν κάποια προβλήματα όσον αφορά την ερμηνεία της συμφωνίας αποχώρησης. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα ήθελα απλά να πω ότι όσον αφορά την κατάσταση που έχει σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς αυτό, αλλά υπάρχουν κάποιοι όροι που είναι αμφίσιμοι, ε, δηλαδή τι ισχύει πριν από το τέλος της μεταβατικής περίοδου ή ε, ποιες ακριβώς είναι διατάξεις που αφορούν στη δικαιοδοσία. Και ως προς την ε, ως προς την ερμηνεία, αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα άρθρα 66-69 τη Συμφωνίας Αποχώρησης, αυτά θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ένωσης θα είναι αρμόδιο για την ερμηνεία Τη συμφωνία, αλλά οι αποφάσει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν θα είναι πλέον δεσμευτικέ για τα Βρετανικά δικαστήρια και αυτά δεν θα μπορούν να ζητούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να τοποθετείται για ασφαλιστικά μέτρα ή για οτιδήποτε παρεμφερέ. Στην περίπτωση τώρα που δεν υπάρξει συμφωνία από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συνάδελφό μου θα πει τι θα κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα έχουμε νομοθετικά εργαλεία, μόνο ένα σημείωμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εδόθη στι αρχές αυτού του έτου και παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο πριν από δύο εβδομάδες. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όσον αφορά το σημείο με αυτό. Να επισημάνω όμως μόνο δύο πράγματα. Όσον αφορά τι διαδικασίε τη συνεργασία σε περίπτωση απαγωγής παιδιού ή συνεργασία για να εντοπιστεί ένα οφειλέτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι ενωσιακοί κανονισμοί δεν θα ισχύουν πλέον, αλλά μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχεια με βάση τη συνθήκη της Χάγης. Ε, βεβαίως αυτό μπορεί να ισχύει αλλά η εμβέλεια αυτών των αποφάσεων της Χάγης δεν είναι ακριβώς η ίδια με τις ενωσιακές αποφάσεις. Μιλάμε για ένα σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο δεν είναι ε, δεσμευτικό, άρα τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν διαφορετικά και μάλιστα τα κράτη-μέλη έχουν ήδη τοποθετηθεί διαφορετικά επ' αυτού του θέματος. Τώρα από την ε, σκοπιά του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δύσκολο να μην παρατηρήσει κανείς ε, την πυρετόδη ατμόσφαιρα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό και δεν θα υπερέβαλε κανείς. Είναι τεράστιο το ποσοστό της απογοήτευσης, 40% και από τις δύο πλευρές υπέρ του Remain και του Brexit ε, αισθάνονται ότι, αισθάνονται ότι δεν πρόκειται να καταφέρουν τίποτα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή που πριν να βγει το Ηνωμένο Βασίλειο, όπω ξέρετε το Βρετανικό Κοινοβούλιο ψήφισε τέσσερι φορέ για το θέμα τη αποχώρηση ε, και τι δύο φορέ που προτάθηκε κάποια συμφωνία ιτήθηκε η κυβέρνηση και υπάρχει και άλλη μια τρίτη ψηφοφορία που μπορεί ή μπορεί να μην οργανωθεί για αυτή την εβδομάδα. Τρεις, τρία συγκεκριμένα είναι τα προβλήματα, πρώτα απ' όλα από την σκοπιά του οικογενειακού δικαίου και είναι προβλήματα με τεράστιες συνέπειε. Πρώτον, τα διαζύγια αυτά καθεαυτά. Το δεύτερον, ε, τα χρήματα που σχετίζονται με τα διαζύγια και μετά η κυδαιμονία των παιδιών, η επιμέλεια. Πράγμα που το υπενήχθηκε προηγουμένω. Ω προ το διαζύγιο το ίδιο, ε, το θέμα είναι ότι αν ε, πρόκειται για διαζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή του Βρετανικού και καθώ θα είναι πλέον ξεχωριστή δικαιοδοσία του Ηνωμένο Βασίλειο, τι θα γίνει με ένα διαζύγιο τη Σκωτία. Θα αναγνωρίζεται στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Και στο βαθμό που δεν θα αναγνωρίζεται, υπάρχει θέμα προτεραιότητας. Ποια ε, διαδικασία ε, διάλυσης ενός γάμου, μιας γαμικής σχέσης θα θεωρείτε ότι υπερισχύει και ποια θα είναι η διαρκής απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου σε τέτοια είδους ε, περιπτώσεις και υποθέσεις. Ποια θα είναι η κατάλληλη δικαιοδοσία και ποιος θα αποφασίζει, ο δικαστής, θα είναι η Lex Pendens που εφαρμόζεται τα τελευταία 25 χρόνια βάσει του ευρωπαϊκού μοντέλου. Επίσης, έχουμε τεράστια, ε, τεράστιο ασφαλιστικά μέτρα, ώστε τα διάφορα μέρη, οι διάδικοι, να μην μπορούν να εκινήσουν άλλη υπόθεση διάλυσης της γαμικής σχέσης, υπόθεση διαζυγίου δηλαδή, στη Γαλλία, στη Γερμανία π.χ. Τι θα κάνει όμως με μια βρετανική απόφαση το ε, άλλο δικαστήριο της άλλης χώρας και πώς θα εφαρμόζεται στην ξένη δικαιοδοσία η απόφαση αναστολής της άλλης υπόθεσης. Θα υπάρχουν λοιπόν δύο ξεχωριστές διαδικασίες για την διαδικασία. Διαφορετικοί δικηγόροι, διαφορετικές δικαστήριων υποθέσεων θα είναι καταστροφικές οι συνέπειες για τα παιδιά. Και αυτό είναι απλώς το πρόβλημα των διαζυγίων. Ε, μέχρι να φτάσουμε να αποφασίσουμε ποιο θα είναι το τελικό η τελική έκβαση του διαζυγίου, τι θα γίνει με τις διατροφές και τα παιδιά. Η διατροφή που είναι ένα βασικό χρηματικό πρόβλημα εδώ. Προφανώς υπάρχει η σύμβαση της Χάγης, όμως δεν είναι ξεκάθαρα το τι συμβαίνει με την δικαιοδοσία. Και εξωτερικός και εσωτερικός στο επίπεδο του καθου κράτους. Και οριζοντίος. Εξωτερικός δηλαδή μεταξύ των διαφόρων συμβαλόμενων μερών της Σύμβασης της Χάγης οι απαιτήσει περί δικαιοδοσίας θα είναι διαφορετικές. Και το τρίτο ε, θέμα, μια πραγματική ρολογιακή βόμβα που θα σκάσει αργά γρήγορα, είναι αυτό των παιδιών. Τι θα γίνει με την συνενετική μεταφορά των παιδιών διασυνοριακά. Το τωρινό σύστημα επιτρέπει στο δικαστήριο τη χώρα ε, παραμονή του να τα κρατήσει στη δικαιοδοσία αυτή για τρει μήνε σε, σε περίπτωση απουσία συμφωνία. Αλλά υπάρχει και το θέμα τη μη συνενετική μεταφορά των παιδιών ε, από τα, μεταξύ των κρατών. Άρα απαγωγή. Η σύμβαση τη Χάγη υποχρεώνει πολλά κράτη παγκοσμίω να ακολουθήσουν του κανόνε. Όμω το καθεστώ που ισχύει τώρα είναι ο κανονισμό τη Βασιλεία. Με ενισχυμένα άρθρα και κανόνε για αντιμετώπιση των υποθέσεων απαγωγών με τρει τρόπου. Πρώτα απ' όλα με επιτάχυνση τη διαδικασία, μετά με ακρόαση του ίδιου του παιδιού, το προσώπο, και τρίτον με την διασφάλιση ότι η χώρα παραμονής έχει δικαίωμα να αναλάβει την ευθύνη ε, της άσκησης πίεσης όταν ε, μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνείται να επιστρέψει το παιδί. Ο λόγος και πάλι στην ε, Μαριέλ. Ναι, στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασης, το τι θα γίνει στο μέλλον και ποιες είναι οι δυνατότητες επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπ' αυτήν την ε, οπτική γωνία, το έγγραφο που έχουμε τώρα είναι η πολιτική δήλωση που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο πέρσι. Εδώ πρέπει να δούμε τι θα κάνει η ομάδα εργασία για θέματα συνεργασία ε, στο αστικό δίκαιο με την κυκλοφορία των πολιτών και τι θα γίνει με την ε, μνήα ε, των συμβαλόμενων μερών πρέπει να επιβεβαιώσουν τη δεσμευσή του στα εργαλεία οικογενειακού δικαίου στα οποία έχουν συμβληθεί, δηλαδή την Σύμβαση τη Χάγη, και να κοιτάξουν κατά πόσο υπάρχουν δυνατότητε δικαστική συνεργασία σε θέματα γαμική ευθύνη και άλλα ε, παρόμοια νομοθετικά θέματα, όπω τι διατροφέ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία δηλαδή όχι μελλοντική συμφωνία, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν κάποιες ε, λύσεις ε, προσωρινές, όπως η Σύμβαση της Χάγης, η οποία όμως δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη. Λόγου χάρη, ε, επειδή το 1970 η απόφαση για τις αναγνωρίσεις διαζυγίων μεταξύ των 100 μελών ε, δεν λύνονται τα προβλήματα. Το ίδιο και το 1973 για την επίλυση των ε, διαφορών ε, διατροφή. Μετά το 1980 δεσμεύονται τα ελακτρωτή μέλη, αλλά παρόλο που τα μέτρα είναι πιο εξελιγμένα, με τον κανονισμό των Βρυξελών 2α τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα, αλλά Εκεί βελτιώνεται μόνο λίγο η θέση των παιδιών. Μετά η διατήρηση των υποχρέσεων διατροφή είναι ακόμα πρόβλημα. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει συμβληθεί στη Σύμβαση αυτή παρόλο που περιμένουν να ξεκινήσει γρήγορα. Ε, εδώ πέρα λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το πεδίο εφαρμογής που ε, έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις ε, διατροφής. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνάψουν ενδεχομένω διμερείς συμφωνίες και δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος επίλυσης γιατί υπάρχει ο κανονισμός του Συμβουλίου ο οποίος προβλέπει μια διαδικασία για τα κράτη-μέλη ώστε να μπορέσουν να συνάψουν διμερείς συμβάσεις αλλά πρέπει να το εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπα και πριν ότι δεν θα μιλήσω πολιτικά, δεν ανήκω ή τέλο πάντων ε, δεν μιλώ ως ε, ε, προσκύμενο σε κάποιο κόμμα. Βέβαια δεν μπορεί κανείς εύκολα να αποφύγει το να μιλήσει πολιτικά με μικρό πι δηλαδή, γιατί μιλάμε για πολίτες. Με πολίτες έχουμε να κάνουμε, πολίτες και των 28 χωρών και με τα παιδιά τους. αυτήν την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και πρόκειται για καταστροφή πραγματική για το οικογενειακό δίκαιο. Και θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι καταστροφή από πλευράς οικογενειακού δικαίου. Υπό την έννοια ότι έτσι όπω έχει η κατάσταση δεν υπάρχει ούτε ένα πλεονέκτημα για του καταναλωτέ. και θα έλεγα ότι υπάρχουν και κίνδυνοι και πολλές ε, ε, παράμετροι που δεν γνωρίζουμε. Και είναι επίγον λοιπόν μέχρι την επόμενη εβδομάδα να λύσουμε τα προβλήματα. Γιατί εδώ μιλάμε για τα παιδιά μας, τα παιδιά και από τις 28 χώρες. Οι επιπτώσεις αυτές από το επόμενο Σάββατο και μετά έχουν να κάνουν με τη βελτιωμένη προστασία, ενισχυμένη προστασία για τα παιδιά, δυνάμει των Βερξελών 2. Μια επιστροφή αρπαγέντων παιδιών και να σας δώσω και ένα παράδειγμα, την πολωνική ε, υπόθεση ενός περιφερειακού δικαστηρίου σε πρώτη και δεύτερη βαθμό MS ε, κατά IS. Ε, Ο λόγος για την άρνηση της μεταφοράς παιδιού ήταν το Brexit και πολιτική αβεβαιότητα, μεταξύ άλλων. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν και στην έφεση και στην πρωτοβάθμια απόφαση του δικαστηρίου και αυτό είναι πρωτοφανές στην ομολογία. Ε, εκεί βλέπουμε την DJ κατά εμέσα ε, που είναι μια άλλη περίπτωση ε, αντίστοιχη μεταξύ Πολωνίας και ε, Αγγλίας εδώ η μεταφορά του παιδιού ε, είναι κράτη μέλη που είναι στα σύνορα και εκεί βλέπουμε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το ενδεχόμενο να υπάρξει μεταφορά παιδιού από το ένα κράτος στο άλλο και ο γονέας που θα μείνει πίσω ε, θα πρέπει να πάει στο άλλο κράτος ε, και να ζητήσει ένδικα μέσα και να προσφύγει με δικά του έξοδα στο άλλο κράτος αυτό ακριβώς γιατί δεν θα εμπίπτει πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και αυτό είναι ο λόγος ε, για τον οποίο πραγματικά η κατάσταση είναι κατεπίγουσα και επικίνδυνη για τα παιδιά όλων των οικογενειών μας. Αυτά είχαμε να πούμε. Ε, σας ευχαριστούμε, κυρία Ρεκέχο, η Σίδρο. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ελπίζω να σας άκουσε κάποιος από το Βρετανικό Κοινοβούλιο μέσω του web streaming. Θέλει κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γιούρη που ανέθεσε την πολύ σημαντική αυτή μελέτη. Την έχουμε μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά και συμφωνούμε ότι στον τομέα του γενιακού δικαίου Έχουμε να κάνουμε με κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά και τις οικογένειές τους από όλη την Ευρώπη. Σε περίπτωση μη συμφωνίας, όπως υπόθηκε, υπάρχουν προβλήματα. Και εμείς έχουμε δώσει ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές με, μια, ένα σημείωμα ετοιμότητας που το παρουσιάσαμε στις 18 Ιανουαρίου και εδώ στην Επιτροπή στις 4 Μαρτίου. Βέβαια, για να έχουμε ασφάλεια δικαίωμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πρέπει να επικυρωθεί το σχέδιο συμφωνίας αποχώρησης. Αυτή είναι η καλύτερη ε, λύση. Υπάρχουν και άλλες ε, επιλογές εναλλακτικέ, αναφέρθηκαν κάποιες, όμως θέλω να πω ότι δεν μιλάμε μόνο για διεθνείς συμβάσεις ε, που αποτελεί μια εναλλακτική, γιατί υπάρχει το εθνικό δίκαιο, αλλά Έχουμε αυτή δηλαδή την εναλλακτική για το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους ή τη διεθνή συμβάση. Ο κ. Σάμο, να απαντήσω αν μου επιτρέπετε. Το εθνικό δίκαιο, ναι, πράγματι συνεχίζει να ισχύει, όμως το μείζον ερώτημα είναι αν υπάρχει μια διαταγή, ας πούμε, στην Αγγλία, πώς θα επιδοθεί σε κάποιο άλλο κράτος ε, στην Ένωση και πώς θα εκτελεστεί. Εκεί είναι το ζήτημα, εκεί είναι το πρόβλημα. Για τα τελευταία 20 χρόνια το πρόβλημα αυτό το έλυναν ε, οι κανονισμοί των Βρυξελών. Αυτό το πλαίσιο. Αν όμως βγει από αυτό το πλαίσιο το νόμενο βασίλειο, κάτι που αναμένεται να συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία το επόμενο Σάββατο, τι γίνεται. Να απαντήσω κι εγώ κάτι. Το Εθνικό Δίκαιο δεν προβλέπει αμοιβαιότητα, λέει η κυρία Γι' αυτό το αναφέραμε κιόλα. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Κυρία και κύριε, και εδώ ολοκληρώνουμε το σημείο 5 και συνεχίζουμε με το σημείο 6. Παρουσίαση των Ευρωπαϊκή Επιτροπών Αποτελεσμάτων ε, τη Διάσκεψη τη Χάγη ε, για τη Σύμβαση για τι Καστικέ Αποφάσει. Στόχος αυτής της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός ε, ομοιόμορφου νομικού πλαισίου για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου. Μια ειδική επιτροπή ε, συστάθηκε το 2016 για την εκπόνηση ενός σχεδίου σύμβασης Εφόσον η αναγνώριση και η τέλεση αποφάσεων είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπεί όλα τα κράτη-μέλη πλην της Δανίας επί τη βάση των οδηγό, οδηγιών διαπραγμάτευσης που ενέκρινε το Συμβούλιο του 2016. Η τέταρτη και η πέμπτη συνάντηση τη ειδική επιτροπή πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018. Οι πρόσωποι τώρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μα ενημερώσουν για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και για τα επόμενα βήματα. Θα παρακαλέσω να περιοριστείτε στα 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon to everybody. Thank you already for introducing the, the, the project. Σας ευχαριστώ Θα ήθελα να αναφέρω τα βασικά στοιχεία της ερευνάς μας. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε τα πορίσματα της έρευνας αυτής. Εδώ θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα της της συνόδου μάλλον για τη σύμβαση τη Χάγης και τα θέματα οικογενειακού δικαίου. Το πρόγραμμα αυτό έχει τις απαρχές του το 1992 και την έγκριση της Σύμβασης της Χάγης, ε, καθώς και την Σύμβαση Επιλογής Δικαιοδοσίας του 1995. για τις δικές αποφάσεις και την ε, επιβολή αυτών στο συγκεκριμένο επίπεδο δικαίου. Όπως είπα, η δουλειά μας ξεκίνησε το 2012. Πολλές ειδικέ επιτροπές ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό και η τελευταία συνεδρία Συνδικής Επιτροπής ήταν το 2008 με ένα σχέδιο κειμένου το οποίο υποβλήθηκε στην Κορεπέρ προς έγκριση. Και η τελική έγκριση του προγράμματος θα γίνει τον Ιούνιο Φέτος, για τις βασικές πτυχές της σύμβασης, πρέπει να πω ότι ένας από τους στόχους είναι να ενισχυθεί πρακτική πρόσβαση στις ε, ε, εκδικάσεις των υποθέσεων και την επιβολή των αποφάσεων, να βελτιωθεί η εμπορική δραστηριότητα με περισσότερη νομική βεβαιότητα, να μειωθεί το κόστος και οι ανασφάλειες. Όλα αυτά για τι διασυνοριακές διαφορές. όπω ξέρετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται... Στι νομικέ διαφορέ λοιπόν αυτού του είδου λείπει ακόμα νομική βεβαιότητα. Υπάρχουν βέβαια περιφερειακέ ε, συμφωνίε όπω η Σύμβαση του Λουγκάνου. της οποίας όμως είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο εφαρμογής. Προκειμένου να καλύψουμε λοιπόν τις έλλειψεις αυτού του, πολυεπί... του πολυμερού επίπεδου συνεννόηση και εφαρμογής τη ε, Σύμβαση τη Χάγη είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σύντομα. Όπω είπατε, Η σύμβαση είναι μεταξύ των αποκλειστικών εξωτερικών αρμοδιότητων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να την εγκρίνει. Εκ μέρους των κρατών μελών με την εξαίρεση της Δανίας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι το τωρινό κείμενο της σύμβασης δείχνει ότι οι υπάρχουσες συνθήκες δεν θα επηρεαστούν από τη νέα σύμβαση. Κατά την άποψή μας, το σχέδιο της ε, κειμένου της σύμβασης προασπίζεται τα ευρωπαϊκά συμφέροντα όπως ορίστηκαν από τις ε, οδηγίες για τις διαπραγματεύσεις. Και προφανώς όλες οι διατάξεις του σχεδίου κειμένου μπορούν να συζητηθούν περαιτέρω. Νομίζω τίποτα δεν είναι αποτυπωμένο σε πέτρα τα βασικά χαρακτηριστικά της σύμβασης που έχουν ως τώρα συμφωνηθεί στο επίπεδο των ε, ειδικών επιτροπών δεν είναι το ίδιο. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν της σύμβασης. Βασικές υποχρεώσεις για να αναγνωριστούν και να επιβληθούν αποφάσεις από άλλα συμβαλόμενα μέρη, ευνοϊκότερη αναγνώριση και επιβολή των δικαστικών αποφάσεων και της εθνικής νομοθεσίας, η σύμβαση θα ισχύει και για εμπορικές διαφορές με ρητή εξαίρεση κάποιων εμπορικών θεμάτων. Στο άρθρο 2 της σύμβασης, ας πούμε, υπάρχει ένας κατάλογος των εξαιρέσεων και μερικά από τα θέματα αυτά εξαιρούνται γιατί ακριβώ καλύπτονται από άλλα διεθνή εργαλεία. Επειδή δεν ισχύει για την διατησία και άλλε σχετικέ ε, διαδικασίε διαμεσολάβηση η σύμβαση, η διατησία θα καλύπτεται από το διεθνέ δίκαιο. Μεταξύ άλλων η σύμβαση της Νέας Υόρκη. Να τονίσω ότι η σύμβαση θα ισχύει για αποφάσεις καταναλωτικών διαφορών ή συμβάσεων εργασίας και θα παρέχει σχετική προστασία τα πιο αδύναμα μέρη, εργαζομένους ας πούμε. Επίσης για τις αποφάσεις και την επιβολή τους. Ό,τι απόφαση και αν πάρει το δικαστήριο θα πρέπει να καλύπτονται οι έξοδικαστικές ε, συμφωνίες και δεν θα καλύπτονται τα θετικά εργαλεία. Θα προβλέπετε ένα σύστημα για την επιβολή ξένων αποφάσεων εάν το δικαστήριο αρχικά πρέπει να βασιστεί σε δικαιοδοσία που καθορίζεται από τη σύμβαση. Εδώ η διάδικοι Θα πρέπει λοιπόν ε, οι ζημίες ε, τιμωρητικού τύπου να καλύπτονται κάπως ε, χρηματικά. Υπάρχει και η σύμβαση των, της Συνεργασίας Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων του 2005 και θα πρέπει το κράτος που υποβάλλει έτοιμα θα πρέπει να επιτρέπει την πρόβλεψη άλλων προστήμων. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τη σύμβαση σκοπεύει να δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο και ε, που να είναι τόσο διαλλακτικό ώστε να εγκριθεί ευρέω στο μέλλον Και παρόμοιο είναι και το πλαίσιο της Σύμβασης της ΧΑΙΣ για την επιλογή των δικαιοδοσιών. Και αν μου επιτρέπετε θα περάσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο, στη συνάδελφο για να σας εξηγήσει σύντομα ποια ζητήματα παραμένουν ακόμη ανοιχτά ή αντιφατικά. Thank you very much and good afternoon. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους σας. Έχουμε ακόμα αρκετό καιρό μέχρι την διπλωματική συνδιάσκεψη και εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα που είναι ανοιχτά. Το πιο σημαντικό είναι ε, κατά πόσον οι διαμάχες ε, για την ε, πνευματική διοκτησία κατά πόσον θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συνθήκη ή όχι. Έχουμε απευθυνθεί στους άμεσους ενδιαφερόμενους πριν από λίγο καιρό και πρέπει να πούμε ότι ενδιαφέρονται μόλις τώρα για αυτή τη συμφωνία που τώρα πια είναι μάλλον πολύ αργά για να γίνουν περαιτέρω διαβουλεύσεις υπάρχουν φόβοι οι οποίοι ίσως ε, να είναι ατεκμηρίωτοι. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν κατά πόσον υπάρχει πρόβλημα με το καθεστώς που ισχύει κυρίως για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα προσέθεται αξία. Υπάρχουν όμως και περισσότεροι φόβοι για το άγνωστο, διότι το ε, ιδιωτικό Διεθνέ δίκαιο είναι ένα πολύ περίπλοκος νομικός τομέα και να εξηγήσει κανείς αυτού τους κανόνες σε ανθρώπους που δεν είναι εμπειρογνώμονες και μερικέ φορές ούτε καν δικηγόροι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Ένα άλλο θέμα που είναι εύκολο να εξηγηστεί είναι ε, πώς ε, τα απλά τα κανονικά δικαστήρια θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συμφωνίας. Αυτά είναι τα δικαστήρια εκείνα τα οποία θα αφορούν δύο περισσότερα κράτη με βάση τη μελλοντική συνθήκη. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είναι common court όπως το αποκαλούμε, κανονικό δικαστήριο όπως το προβλέπει η συμφωνία, γιατί μιλάμε για μια συμφωνία η οποία εμπίπτει στην αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ένα μέρος και το δικό της δικαστήριο είναι αυτό στο Λουξεμβούργο. Αυτό είναι το δικαστήριο του ενός συμβαλόμενου μέρους. Τα κανονικά δικαστήρια είναι πιο σημαντικά στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μιλάμε ε, για το δικαστήριο δικαστήριο που έχει σχέση με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή με το δικαστήριο ε, για τις χώρες ε, Μπενελούξ. Κατόπιν, υπάρχει κι άλλο ένα θέμα το οποίο επ' αυτού δεν συμφωνούμε, είμαστε ακόμα πολύ μακριά, είναι οι αποφάσεις των κυβερνήσεων. Γιατί έχουμε κάποια κράτη ε, στην Τράπεζα Διαπραγματεύσεων που εξακολουθούν να θέλουν να ισχύει πεπατημένοι τη ε, της απόλυτης ε, ασυλίας, ξεπερασμένο αυτό, για αυτούς η δεν εμπίπτει σε αρμοδιότητες ενός κράτους, αλλά η πλειοψηφία των συμβαλωμένων ε, θεωρεί ότι το μόνο που αποκλείεται είναι τα εμπορικά θέματα. Υπάρχουν λοιπόν ε, προσπάθειες να εξαιρείται μόνο το ακτεγιούρια την Πέρια Ένα πράγμα πρέπει να είναι απόλυτα σαφές, ε, δηλαδή οι κρατικές επιχειρήσεις να μην καλύπτονται από αυτές τις εξαιρέσεις, γιατί και αυτές ε, ε, διαπραγματεύονται όπως τα νομικά ή τα φυσικά πρόσωπα και θα πρέπει να εξαιρούνται από τη συμφωνία. Κατόπιν υπάρχει και ένα θέμα σχετικά με την ιδιωτικότητα και τις αποφάσεις ή τις διατάξεις που αφορούν τα τρας, του ομίλου επιχειρήσεων. Πολλοί πιστεύουν ότι όλα αυτά θα πρέπει να αποκλείονται. Και επίσης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας εκεί έχουμε αποφάσεις για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και στις περιπτώσεις αυτές χρειαζόμαστε καλύτερη διατύπωση για να μπορούμε να εκφράσουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το αποτέλεσμα σχετικά με την ισχύ. Ένα άλλο θέμα, και αυτό είναι το τελευταίο που εξακολουθεί να είναι ανοιχτό, είναι το θέμα των διμερών συμφωνιών, δηλαδή όταν ένα νέο κράτος προσχωρεί στη συμφωνία. Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία επιθυμούν να μπορούν να αποφασίζουν σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση ε, κατά πόσον θέλουν να έχουν ε, συμβατικές σχέσεις συμφωνίες με ένα νέο κράτος μέλος. Αυτό ισχύει και για άλλες ε, συμφωνίες της Χάγης. Για μερικούς η ε, σιωπή σημαίνει συνένεση. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο όπου τα κράτη-μέλη μπορούν να εκφράσουν την αντίρρησή τους. Άλλοι λένε πάλι ότι πρέπει να ισχύει ένα διαφορετικό μηχανισμό να εκφράζει κανείς την διαφωνία του με απόλυτη σαφήνεια. Ε, αυτό πρέπει ακόμα να το αναλύσουμε, δεν έχουμε καταλήξει. Όταν συζητήσαμε εδώ την τελευταία φορά, τέθηκε ένα ερώτημα, δηλαδή τι θα γίνει αν ένα κράτος προσεχώρησε και έγινε αποδεκτό. Αργότερα όμως αλλάζει το νομικό σύστημα αυτού του κράτους και δεν γίνεται πλέον σεβαστό το κράτος δικαίου. Εμείς από πλευράς Επιτροπής πιστεύουμε ότι η εξαίρεση της δημόσιας πολιτικής αρκεί για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, αλλά σε πολλές άλλες περιπτώσεις η συνθήκη της Βιέννης επιτρέπει και αυτή να ανασταλεί η συνθήκη της Χάγης σε διμερείς σχέσεις. Αυτά λοιπόν μπορούμε να περιμένουμε ως προς τη διπλωματική διάσκεψη τον Ιούνιο. Και υπάρχει και μία, ένα ερώτημα το τι θα ακολουθήσει μετά. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται το ερώτημα ε, πότε τα κράτη-μέλη θα μπορούν να απευθυνθούν στο δικαστήριο. Ε, συμφωνήσαμε στη Χάγη ότι αυτό θα είναι μια επόμενη διαδικασία και η, επόμενη, και η πρώτη συνάντηση των εμπειρογνωμόνων επί του θέματος θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Έχει ανακοινωθεί. Αυτά είχαμε να σας πούμε και βεβαίως είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δοκιμάζω ένα άλλο μικρόφωνο. Μ' ακούνε οι διερμηνείς, ωραία. Έχετε ερωτήσεις προς τους ε, προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ για την παρουσίαση και έτσι ολοκληρώνουμε και αυτό το σημείο, το σημείο 6 και προχωρούμε στις ψηφοφορίες.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 So, dear Αγαπητοί συνάδελφοι, να προχωρήσουμε με τις ψηφοφορίες. Πρώτη αφορά την νομική βάση για τους καταγγέλλοντες. Ο κύριος Λεμπρετών, ο εισηγητής μας, δεν είναι εδώ. Μήπως έχει πει σε κάποιον από εσάς να τον εκπροσωπήσει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Α, όχι. Δεν έχει ζητήσει κάποιον από κάποιον να διαβάσει κάτι εξ αυτού. Έχουμε από την κυρία Ροζιέρ μια προφορική τροπολογία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Ροζιέρ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, υπάρχει μια προφορική τροπολογία σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για την νομική βάση άρθρο 39 προταστασία ατόμων που καταγγέλνουν παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας. Προτείνουμε τις εξής προφορικές τροπολογίες στο τμήμα 5 ανάλυση και προσδιορισμός τη ενδεδημής νομικής βάσης προτίθεται στην 5 το εξής κείμενο σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι το άρθρο 31 της συνθήκης Ευρατόμα αναφέρεται σε μια διαδικασία μη νομοθετικής φύσεως. Ωστόσο υπάρχουν προηγούμενα τα οποία συνδυάζουν νομοθετικές και μη νομοθετικές διαδικασίες επί παραδείγματι η Οδηγία 2014 κάθος 104 Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Νοεμβρίου 2014 για ορισμένου κανόνες ε, που διέπουν ε, τις, ε, την αποζημίωση δυνάμει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις διατάξεων του νόμου περί των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 103 μη νομοθετικό και 114 νομοθετικό τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τμήμα 6 συμπεράσματα και συστάσεις προτείνεται στο τέλος της δεύτερης παραγράφου το ακόλουθο κύμα δεδομένων των τομέων πολιτικής και των μέτρων που καλύπτονται από το κείμενο ε, δυνάμει της, της προσωρινής συμφωνίας ε, το η νομική βάση ορίζεται ως δι και σταματάει εκεί. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε καταρχάς την προφορική αυτή τροπολογία και εν συνεχεία τη γνωμοδότηση συνολικά. Ελπίζω να έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, αρχίζει ψηφοφορία. One more, maybe. Αφήνω άλλο λίγο χρόνο. πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, μία κατά και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της νομοδότης. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα και συγχαρητήρια στον κύριο Λεμπρετό. Έχουμε μια δεύτερη έκθεση Λεμπρετών, νομική βάση για τα καλυπτόμενα ομόλογα. Άρχεται η ψηφοφορία. Yep, ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται και συγχαρητήρια για μια ακόμη φορά στον κύριο Λεμπρετών. Και τώρα, έκθεση Ροζιέρ. So may I first give the floor to my... Θα ήθελα να δώσω καταρχάς το στην κυρία Ροζιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για την οδηγία για την προστασία των καταγγελόντων το αποτέλεσμα του Κοινοβουλίου είναι σύμφωνο με την εντολή που είχαμε από τη, στη δική μας Επιτροπή. Έχουμε ένα κείμενο που προστατεύει, που παρέχει εχέγγυα, ευελιξία για την προστασία των καταγγελόντων. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων μορφών ε, καταγγελίας εκ μέρους των ανθρώπων αυτών. Έγινε πολύ ομαδική δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κιώδης γιατί μόνιμα ήταν διαθέσιμη ιδίω η κυρία Καβαντά, Ντιράν, ήταν σε όλες τις συναντήσεις ε, και συνέβαλαν και αυτοί στο να έχουμε ένα αποτέλεσμα απόλυτα ευθυγραμμισμένο με αυτό που είχαμε αποφασίσει ως Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Κοινοβούλιο. Είμαστε ομόφωνοι σε ό,τι αφορά την εντολή και ελπίζω το ίδιο αποτέλεσμα να έχουμε ε, και σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα αυτή των ε, διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι για το αποτέλεσμα. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Yes, Πέρας, ομόφωνα δεκτή έκθεση γαριτήρια. Να προχωρήσουμε με το σημείο 9 της μερισιάς διάταξης. Πρόγραμμα δικαιοσύνη. Κυρία Χάουταλα και ο κύριος Βάιντενχόλτσερ ήταν οι εισηγητές. Έχουμε λοιπόν την αναφορά εκ μέρους των από τον εισηγητών, κύριε Χάουταλα, να καλωσορίσω και το συνεισηγητή μου. Ε, συνεδριάζομαι στην Επιτροπή Γιούρη. Αυτό το θέμα έληξε μετά από δύο πολιτικούς τριμερείς διαλόγους και έξι τεχνικές συναντήσεις και μη ιδιαίτερα ευγνώμων στη γραμματεία χάρη στην οποία όλα τα πολιτικά σημεία που είχαμε έγιναν τελικά δεκτά μέσα σε δύο εβδομάδες, μέσα σε δύο συναντήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό και θεωρώ ότι θα πρέπει να το στηρίξουμε. Και εδώ και στην Ολομέλεια το κείμενο γραμμίζεται με το πρόγραμμα δικαιώματα και αξίες που διαπραγματευόμασταν ταυτόχρονα. Ε, το βασικό επίτευγμα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ένα άρθρο 3α νέο για την συμπερίληψη της διάταξης του φύλου και των δικαιωμάτων των παιδιών και τη μη τεκτική μεταχείριση. Ό,τι δηλαδή περιλαμβάνει το άρθρο 21 του χάρτη. Εμείς επιμείναμε και πετύχαμε η προοπτική της ε, ισότητας των φύλων να περιλαμβάνεται στους δείκτες παρακολούθησης του προγράμματος. Επίσης, η ανεξάρτητη αμεροληψία του δικαστικού σώματος και ο ρόλος για την ενίσχυση της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου των δικαιωμάτων αναφέρονται με μεγαλύτερη έμφαση, αν και το Συμβούλιο ήταν κάπως διστακτικό και έπρεπε να τους υπενθυμίζουμε ότι το κράτος δικαίου και οι ευρωπαϊκές αξίες ε, πρέπει να περιλαμβάνονται παντού και όχι μόνο σε αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, το παράρτημα στο οποίο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες του προγράμματος ε, περιλαμβάνει παράγραφο για τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ο συνεισηγητής μου θα το τονίσει φαντάζομαι με τη σειρά του. Ήταν σημαντικό και για τους δυο μας αυτό. Τώρα λοιπόν έχουμε την σχετική παράγραφο στο κείμενο. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και στα επόμενα βήματα. Μιλάμε για το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο, γιατί εκεί εντάσσεται αυτή, αυτό το πρόγραμμα. Η διαδικασία δεν είναι ξεκάθαρη. Περιμένουμε επιστολή από το Συμβούλιο, όπου θα διευκρινίζει τις θέσεις του το Συμβούλιο, διότι αυτή τη στιγμή η έκβαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων είναι μια μερική προσωρινή συμφωνία, μια προσέγγιση που επελέγει διότι δεν έχει εντολή το Συμβούλιο για πλήρης διαπραγματεύσεις, μόνο για κάποια στοιχεία, τα περισσότερα από τα οποία ε, αφορούν τα νούμερα, τα συγκεκριμένα, μπήκαν σε αγγύλες και άρα δεν μπορούσαμε να τα διαπραγματευτούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα συνολικό ζήτημα που αφορά όλες τις επιτροπές του Κοινοβουλίου και η διατύπωση που χρησιμοποιείται είναι ότι το, η έκβαση των διαπραγματευτών αποτελεί την κοινή συνεννόηση των διαπραγματευτών. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να αναγνωριστεί νομικά η όρος, δηλαδή κοινή συνεννόηση, που είναι και με την επιφύλαξη της τελικής έκβασης ε, των διαπραγματεύσεων, του πλήρους κειμένου δηλαδή. Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να επαναληφθούν μόνο όταν θα έχει το Συμβούλιο πλήρη εντολή, που σημαίνει την επόμενη θητεία. Όσο λοιπόν ε, και αν θεωρώ ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε πλήρως αυτή την κοινή συνεννόηση που έχει επιτευχθεί, θα πρέπει να δούμε τελικά το Συμβούλιο πώς ε, ε, θα δείξει στην πράξη τι αντιλαμβάνεται με αυτή την κοινή συνεννόηση. Έχουμε κάποια συμπεφωνημένα σημεία τα οποία δεν θα πρέπει να ξανανοίξουν στο πλαίσιο της συμφωνίας. Θα δούμε τη δέσμευση του Συμβουλίου σε αυτό. Τον τρόπο, το μοναδικό τον πρωτόγνωρο διαδικασία. Επίσης, για την κοινή αυτή συνόηση, την Πέμπτη η το πρωί θα ψηφίσουμε σε μια κοινή συνεδρίαση Γιούρι Λίμπε. Η διάσκεψη των Προέδρων όμω μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιώσει ακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα διαδικαστικά βήματα ε, στο Κοινοβούλιο. Περιμένω λοιπόν την Πέμπτη στην Επιτροπή Γιούρη και Λίμπε να ψηφίσουμε και να επιβεβαιώσουμε τη θέση της, ε, του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, όπως πρέπει την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Δεν ξέρουμε τώρα ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου για αυτή την κοινή συνεννόηση. Δεν έχουμε από τη διάσκεψη των Πρόεδρων επίση κάποιο νεότερο, άρα ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγέ. Και αν πράγματι συμβεί αυτό, είμαι βέβαιη ότι και η Γραμματεία, αλλά και εμεί βέβαια οι συνεισηγητέ θα σα ενημερώσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε θέλετε Συμφωνώ πλήρως με, με την εισηγητρία. Άλλα σχόλια από, τα, από σας, από κάποιον άλλον, από ό,τι φαίνεται όχι. ω εκ τούτου συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 10. Είναι η αναφορά στην Επιτροπή ε, σχετικά ε, με τις ε, μετατροπέ, μετατροπές. Ε, η κυρία Ρίγνερ νομίζω. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και χαίρομαι που μου προσφέρετε αυτή η ευκαιρία να σας ε, ενημερώσω εκ μέρους της ε, εισηγήτριας της κυρίας Ρέγνε σχετικά με το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις ε, που εντάσσονται στο εταιρικό δίκαιο. Η συμφωνία κατέληξαν οι συνομοθέτε στο Στρασβούργο από αυτού του θέματος και η εισηγήτρια θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους, κυρίως τους και οδηγητές, ε, τους συνεργάτες τους και τις υπόλοιπες ομάδες των άλλων ε, θεσμών για την πάρα πολύ καλή δουλειά, μια επικοδομητική προσέγγιση για να εξευρεθεί συμφωνία. Έτσι λοιπόν ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η δουλειά του να ε, συμφωνήσουμε όλοι πάνω σε αυτή την ιδιαίτερα επίμαχη το επίμαχο θέμα. Κάποια στοιχεία της μελλοντική οδηγίας είναι ότι η Κορεπέρ θα εγκρίνει το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου στις 27 Μαρτίου. Και η ψηφοφορία στη Γιούρη θα λάβει χώρα ε, την 1η και τη 2η και στις 2 Απριλίου του 19 και οι δύο οδηγίε ε, του πακέτου εταιρικού δικαίου ε, θα παραμείνουν ενωμένε, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν τον Απρίλιο στο Στρασβούργο. Γιατί γι' αυτό είχαμε ασκήσει πίεση. Η οδηγία ε, προβλέπει μία εναρμονισμένη ενιαία διαδικασία και για τις τρεις αυτές εταιρικέ διαδικασίες, τις μετατροπές, τις συγχωνεύσεις και τις διαιρέσεις. Μετά από την ε, προσέγγιση και παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένουν οι ίδιες ε, δικλείδες ασφαλείας και για τα τρία θέματα της εταιρική κινητικότητας. Και έτσι θα καταστεί δυνατόν να υπάρχει διαιτησία και κάποια ασφάλεια για τις αρμόδιες εθνικές αρχές και για τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Οι νέοι κανόνες για την εταιρική κινητικότητα ε, προσφέρουν στις τίμιες εταιρείε νέες διαδικασίες, οποτεδήποτε επιθυμούν ε, διασυνοριακά να προβαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες και διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη ορίζουν μια αρμόδια υπηρεσία η οποία ορίζει μία και μόνο εφαρμογή και για τις ε, συγχωνεύσεις και για τις ιερέσεις και οποτεδήποτε ζητηθεί ένα σχετικό πιστοποιητικό. Ε, η βασική εξουσία ε, αποδίδεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, το να υπάρχει το, η απέτηση να υπάρχει ένας ε, ανεξάρτητος ε, νομικός εμπειρογνώμονας. Ε, αυτός έχει απλά ένα λογιστικό ρόλο. Η έκθεση στα μέλη και στους υπαλλήλους προβλέπει μία και μόνο έκθεση και διατηρούνται βασικά στοιχεία της έκθεσης. Η αρμόδια αρχή τα λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ε, διασυνοριακές ε, διαδικασίες ε, ως προς τις μετατροπές, τις συγχωνεύσεις και τις διαιρέσεις. Όσον αφορά τώρα τους όρους, αυτοί θα κοινοποιηθούν και εκεί προβλέπεται καλύτερη ενημέρωση για τις θηγατρικές εταιρείες, για κίνητρα. Η εταιρεία λοιπόν πέντε χρόνια πριν από τη διασυνοριακή ε, αυτή δράση θα πρέπει να έχει λάβει όλες τις ε, απαραίτητες ε, πληροφορίες και θα πρέπει να υπάρχει και ένας έξτρα κατάλογος πληροφοριών που θα κατατίθεται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή. Ε, η συνεργασία με άλλες αρχές, τα κράτη-μέλη, αυτή θα ενισχυθεί έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη διασυνοριακή ε, δράση. Εξάλλου, η αρμόδια αρχή ε, θα πρέπει να ενημερώνει κυρίως στο κράτος μέλος το οποίο έχει ενδιαφέρον στο να παραμείνει εταιρεία, να καταβάλει όλους τους φόρους, να προστατεύει τους εργαζόμενους πριν ε, χορηγηθεί ε, το πιστοποιητικό για την διασυνοριακή ε, μετακίνηση. Και στα τρία αυτά κεφάλαια προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας κατά του ενδεχόμενου των καταχρήσεων. Η αρμόδια αρχή δεν θα εκδίδει το απαραίτητο πιστοποιητικό αν ε, μέσα από την αξιολόγηση των διαδικασιών της, διαδικασιών της εταιρεία διαπιστώσει ότι η δράση αυτή θα γίνει για, ε, με στόχο την απάτη, την κατάχρηση ή αν θέλετε και την ε, αποφυγή, παράκαμψη του δικαίου και του ενωσιακού δικαίου. Γίνεται αυτή η διαδικασία για να μην καταβληθούν μισθοί και παρεμφερεί. το να, ε, για να μπορεί η αρμόδια αρχή να έχει κάποια καθοδήγηση, οι συνομοθέτες συμφώνησαν να υπάρχει ένας μη εξαντλητικός κατάλογος παραγόντων όπως τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ή της μονάδας στο κράτος μέλος όπου ε, θα καταγραφεί η εταιρεία μετά την διασυνοριακή δράση. Το περιεχόμενο ε, του εγχειρήματος ε, το, ο καθαρός κύκλος εργασιών, ο αριθμός των υπαλλήλων, η σύνθεση του ισολογισμού, τα κεφάλαια, ο εξοπλισμός Επίσης θα πρέπει να καταγράφεται ο χώρος εργασίας των εργαζομένων μιας ε, συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων. Να καταγράφεται και ο αριθμός ε, ε, των εργαζομένων σε μια άλλη χώρα να καταγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν αποσπαστεί τη χρονιά πριν από το εγχείρημα ε, και ο αριθμός εργαζομένων που έχουν καταγραφεί την ίδια στιγμή σε περισσότερα κράτη-μέλη. Επίσης, να καταγράφεται και το που πρέπει να καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έχει ε, τεκμηριωμένες υποψίες για κατάξη, μπορεί όλη, όλο το εγχείρημα να επεκταθεί ε, σε τρεις κατά τρεις περαιτέρω μήνες. Η κυρία Ρέγνε λέει ότι με όλες αυτές τις ε, διαδικασίες. παρόλα αυτά πρέπει να υπάρχει πλήρης ε, σεβασμός ε, του κεκτημένου να ενταχθεί και ένα ξεχωριστό άρθρο ε, σχετικά με την ενημέρωση και στα ε, τρία διαφορετικά κεφάλαια. Εκεί θα υπενθυμίζεται το χρονικό πλαίσιο που πρέπει να ισχύει για την ενημέρωση και τις διαβουλεύσεις. Οι συνομοθέτες διευκρίνησαν ότι όχι μόνο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων αλλά και τα εργασιακά ε, συμβούλια όλοι αυτοί θα πρέπει να ενημερώνονται και να ε, ζητείτε η γνώμη τους. Όσον αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων, στον τελικό τριμερή ε, διάλογο οι συνομοθέτες συμφώνησαν να συμμετέχουν καλύτερα οι εργαζόμενοι. Το Συμβούλιο δέχτηκε ε, να ορίσει ένα όριο και στις τρεις αυτές διαδικασίες προκαλώντας βέβαια τις ε, διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους από τη στιγμή που μία επιχείρηση έχει ε, ξεπεράσει το ανώτατο όριο. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόρθωσε να επεκτείνει ε, το χρονικό διάστημα εφαρμογής από τρία σε τέσσερα χρόνια. Τέλος, το Κοινοβούλιο επίσης κατόρθωσε να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία σε περιπτώσεις όπου μια εταιρεία μεγαλώνει ε, με διασυνοριακές δράσεις και ε, το όριο το φτάνει μόνο μετά τη μετακίνηση. Αυτό είναι απαραίτητο για να υπάρχει ε, μια εναρμόνιση και Τώρα λοιπόν το καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σκεφτεί πότε θα προβεί σε αναθεώρηση αυτής της οδηγίας. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι οι συνομοθέτες μπόρεσαν να βελτιώσουν την διαφάνεια και να συμφωνήσουν ε, σε ελέγχους σε ένα άρθρο που προβλέπει ότι εάν υπάρχει δόλος ή απάτη, αν εντοπιστεί αυτό μόνο μετά τις ε, διασυνοριακές δράσεις, τότε οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν ε, να επιβάλλουν αναλογικά πρόστιμα. Ήταν ένα πολύ μακρύ μήνυμα από την εισηγήτρια για μια πάρα πολύ σημαντική οδηγία. Δεν ξέρω αν έχουν ερωτήσεις οι βουλευτές, από ό,τι βλέπω όχι. Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο υπαριθμών 12 που είναι η, ε, τα πιστοποιητικά προέλευσης και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, στην κυρία Ροζιέρ. Δηλαδή εμένα. Την περασμένη εβδομάδα το κείμενο αυτό που σκοπό έχει να διασφαλίσει την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, πράξη τη Γενέβη, δηλαδή ένα διεθνέ σύστημα αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων, είχαμε δύο τριμερεί διαλόγου. Στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα στι 11 και στι 13 του μήνα. Ο πρώτο ε, εισαγωγική προετοιμασία και ο δεύτερο ολοκλήρωση του θέματο. Πολύ γρήγορα από για το πράγμα. Ε, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, πρέπει να τους ευχαριστήσουμε εδώ, έδειξαν πολύ καλή διάθεση να ικανοποιήσουν ε, τις δικέ μα απαιτήσει. και έτσι μπορέσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Κάτι μόνο μας απογοήτευσε, το είχαμε υπογραμμίσει ω προ τη θέση μα γενικότερα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να προσχωρήσει ε, απολύτως στην ε, πράξη της Γενέβης γιατί εκεί προστατεύονται οι γεωργικές και μη γεωργικές ονομασίες εκεί όμως που δεν ε, εμείς έχουμε νομοθεσία είναι για τις μη γεωργικές ενδείξεις οπότε εκεί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλήρως την πράξη της Γενέβης τώρα η ρήτρα αναθεώρησης που επίσης περιλαμβάνεται στο κείμενο δίνει τη δυνατότητα εντελεχούς ανάλυσης εφόσον χρειαστεί των ελλείψεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ώστε να μπορέσουμε πλήρως να αξιοποιήσουμε αυτή την πράξη της Γενέβης και μελλοντικά να δούμε τη δυνατότητα να καλυφθούν και οι γεωγραφικές ενδείξεις μη γεωργικού χαρακτήρα. Επίσης, ε, οι τροπολογίες που έγιναν στο αρχικό κείμενο, ε, ε, κατάλογο δηλαδή των γεωγραφικών ενδείξεων, θα περιληφθούν στο διεθνές σύστημα που σκοπό έχει να λάβει υπόψη τις απαιτήσεις των οικονομικών φορέων. Ένα εργαλείο που σκοπό έχει να προστατεύσει τους παραγωγούς, να τους δώσει το λόγο για να μπορέσουν και οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες των διατάξεων. Και επειδή δεν προστατεύονται οι γεωγραφικέ ενδείξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση που μπορεί να προκύψει και που ελπίζουμε να είναι προσωρινή μόνο για τα περισσότερα κράτη-μέλη, που έχουν όμω εθνική προστασία για τις μη, γεωγραφικές, για τις μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις και τις έχουν καταγράψει στο προηγούμενο διεθνέ σύστημα, αλλά με την συμφωνία της Λισαβόνας επιτρέπεται η γεωγραφική ένδειξη να προστατεύεται. Κάποιοι λοιπόν έχουν καταχωρημένες τις προστασίες τους στο παλιό σύστημα, έπρεπε λοιπόν να δούμε μια μεταβατική λύση. για να μπορέσουν να λειτουργούν εκ, του, εκ και τα δύο συστήματα, το παλιό και το καινούριο. Η συμφωνία είναι καλή. Θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην πράξη τη Γενέβη για τι ονομασίε προέλευση και γραφικέ ενδείξει, POP και PIP. Και θα προσπιστούμε την τροπική παραγωγή σε πρώτη φάση γεωργική και κτηνοτροφική για μετά και μη. Στο επίπεδο διεθνού εμπορίου. Είναι θετικότατο. Και για του παραγωγού μα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανεί το λόγο. Έχετε κάτι να προσθέσετε. Όχι. Είναι εδώ ο κύριος Μπέτφορτ από την DG Agri. Παρακαλώ, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Γιούρι και την ομάδα της εισηγήτρια για την φοβερή δουλειά που έγινε στο το σκέφτο και την τεχνική και την καλή συμβαστική σας διάθεση για να βρεθεί γρήγορα μια λύση. Το θέμα είναι ότι όλοι είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τις μη γεωγραφικές, μη γεωγραφικές ενδείξεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε ε, την παράλληλη λειτουργία των δύο συστημάτων, παλιού και καινούργιο, μετά την έγκριση της πράξης της Γενέβης, όπου ζήτησε το Ευρωκοινοβούλιο. Και ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και δήλωση για την ενεξελίξη μελέτη και για τη μελλοντική δυνατότητα προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της καλύτερης νομοθεσίας, της, καλύτερης, ε, της ταχύτερης νομοθεσίας και της πιο εύληπτης, θα ενημερώσουμε λοιπόν σχετικά σύντομα. Και θα δούμε πόσο μπορεί να υπάρξει αυτή η διεύρυνση του πεδίου. Ευχαριστούμε όμως την εισηγητή για τη φοβερή της δουλειά καθώς και την ομάδα της. Ευχαριστώ. Thank you very much. Thereby we can close this point. Uh, Μπορούμε να κλείσουμε αυτό το σημείο. Μπορούμε. Και τα επόμενα σημεία είναι κλεισμένα των θυρών, οπότε θα παρακαλέσω τους μη έχοντες εργασία να αποχωρήσουν. Thank you.